Συνάδελφοι, παρακαλώ καθίστε. Έχετε Γερμανό πρόεδρο προς στιγμή. Προσοχή. Είναι μεγάλη μου χαρά που σας καλωσορίζω στην ε, ε, συνεδρίαση της Επιτροπής μας που θα συσταθεί σε σώμα για να δούμε τις παρανομίες ε, που έχουν να κάνουν με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και την αποφυγή της σε σχέση με, το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, τη φοροαποφυγή και τη φοροδιαφυγή. Θα ονομάζεται ΠΑΝΑ αυτή η Επιτροπή. Ε, Ευτυχώ που μέσα από όλο αυτό το μακρινάρι μπορέσαμε να φτιάξουμε αυτόν τον τίτλο ΠΑΝΑ, για να το καταλαβαίνουν όλοι. Πρώτα απ' όλα κηρύσω την έναρξη τη συνεδρίαση να σα πω ότι σκοπός της συνεδρίασης είναι να εκλέξουμε το Προεδρείο της Επιτροπής και τους Αντιπροέδρους βάσει των άρθρων 191 και 204, 198 και 204 του εσωτερικού κανονισμού. Ε, προβλέπεται πρώτα η εκλογή του Προέδρου και μετά των Αντιπροέδρων. Θα ε, πω ότι οι μόνιμοι και αναπληρωτές που θα, τα τακτικά μέλη και οι αναπληρωτές που θα περιληφθούν στην ψηφοφορία πρέπει να ανακοινωθούν και εφόσον υπάρχουν αλλαγέ από τι διάφορε πολιτικέ ομάδε, πρέπει να ανακοινωθούν στο Προεδρείο πριν γίνει η ψηφοφορία. Για την, για την ώρα δεν έχω καμία τέτοια ένδειξη, οπότε θα προχωρήσω με τον κατάλογο τη ψηφοφορία όπω έχει ανακοινωθεί από τι πολιτικέ ομάδε. Για να επαληθεύσουμε, αν και το έκανα μετρώντα, έχουμε απαρτία. Ένα τέταρτο των μελών. Βλέπω ότι είμαστε πάνω από 17 μέλη της Επιτροπής μας. Οπότε ελπίζω να είναι και πάντα έτσι η προσέλευση. Όπως και σήμερα για την ε, καταστατική μας συνεδρίαση. Να περάσουμε στο σημείο 1 της ημερήσιας διάταξης, εκλογή του Πρόεδρου. Θα ήθελα να ακούσω τι υποψηφιότητε και να πω ότι ο υποψήφιο μπορεί να προταθεί μόνο από πολιτική ομάδα ή από το 5% των μελών τη Επιτροπή. Υπενθύμηση είναι αυτή. Και παρακαλώ να μου κάνετε τις προτάσεις σας. Ο κύριος Ροζάτη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εκ μέρους του ΕΛΚ θέλω να υποβάλω την υποψηφιότητα του συναδέλφου Λάγκεν. Γνωρίζουμε όλοι τον Βέρνερ Λάγκεν. Είναι έμπειρος ευρωβουλευτής είναι στο Ευρωκοινοβούλιο πάνω από 20 χρόνια και ε, συμμετέχει εκτός των άλλων στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων. Έχει μακρά εμπειρία σε θέματα οικονομικά και φορολογικά και νομίζω ότι θα είναι εξαιρετικός υποψήφιος για την Προεδρία αυτής της Επιτροπής, της Εξεταστικής Επιτροπής. Ευχαριστώ πολύ. Έχουμε την υποψηφιότητα του ΕΛΚ, ο κ. Βέρνερ Λάγγεν. θα είναι τακτικό μέλος της Επιτροπής ο κ. Λάγκεν, αλλά τον, ε, θέλω να τον ρωτήσω αν έχει υπογράψει την δήλωση οικονομικών συμφερόντων και αν θέλει να λάβει και ένα τέτοιο βαρύ καθήκον. Κύριε Λάγκεν, ευχαριστώ πολύ για τη στήριξή σας. Κανένα πρόβλημα. Δέχομαι την υποψηφιότητα. Άρα συμπεραίνω ότι και την υποψηφιότητα δέχεστε και έχετε υποβάλει και τη δήλωση οικονομικών ε, στοιχείων. Διαβοής Ελπίζω ότι δέχεστε την υποψηφιότητα, εφόσον δεν υπάρχει άλλο υποψήφιο. Ο κύριος Λάγγεν λοιπόν εκλέγεται πρόεδρος αυτής της επιτροπής και τώρα μπορούμε να ανταλλάξουμε θέσεις. Σα ευχαριστώ. Yes, Ευχαριστώ πολύ για την στήριξή σας. Θα ήθελα να είναι δίκαιη, διαφανής, εύκολη η δουλειά της Επιτροπής Πάνα και αποτελεσματική μέχρι την τελευταία μας, την τελική μας έκθεση. Να περάσω τώρα στη μητρική μου γλώσσα, στα γερμανικά δηλαδή. Έχουμε διερμηνία σε όλες τις γλώσσες από ό,τι βλέπω. Θα ήθελα και στα γερμανικά να σας ευχαριστήσω ένθερμα για την εμπιστοσύνη σας. Είναι πολύ σημαντικό το καθήκον που αναλαμβάνω, γιατί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να δείξει ότι τα θέματα της ε, τα φορολογικά, της φορολογικής δικαιοσύνης. Ε, βεβαίως ε, θα ληφθούν σοβαρά υπόψη και σύμφωνα με την τάξη 1 και τάξη 2 και θα ήθελα να ε, έχουμε καλή και δίκαιη συνεργασία με όλους και με καλά αποτελέσματα βέβαια. Η Εξεταστική Επιτροπή είναι ένα από τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας ώστε και απέναντι στα κρατημέλη αλλά και απέναντι στους άλλους ε, θεσμικούς, ε, στα άλλα θεσμικά όργανα να καταστήσουμε αυτή τη θέση μας. Εγώ ε, χαίρομαι που θα έχουμε πολύ καλή συνεργασία με όλους τους συναδέλφους και με τους συντονιστές και τώρα καλό είναι να περάσουμε στην εκλογή του Αντιπροέδρου έτσι ώστε στο τέλος αυτής της 11μηνης εντολής να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε καλά αποτελέσματα. Και πάλι σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την στήριξή σας. Πάμε λοιπόν στην μέση διάδεξη. Σημείο 2. Εκλογή των αντιπροέδρων. Στην απόφαση της Ολομέλειας καταγράφεται ότι η Επιτροπή θα εκλέξει τέσσερις α, αντιπροέδρους. Έχουμε προτάσεις, έχουμε υποψηφίους. Καταρχάς να ρωτήσω αν υπάρχουν άλλες επιθυμίες πριν περάσουμε κατευθείαν στην ψηφοφορία. Υπάρχουν, υπάρχει κάποιος που να θέλει το λόγο. Από ό,τι βλέπω όχι. Οπότε, περνούμε στον πρώτο υποψήφιο, πρώτο αντιπρόεδρο. Υπάρχει συμφωνία της Γενικής Γραμματείας, την οποία έχω στα χέρια μου, όπου ο πρώτος αντιπρόεδρος θα είναι από τους ε, Δημοκράτες και Σοσιαλιστές, από το S&D. Παρακαλώ λοιπόν τις προτάσεις σας. Ο κύριος Σίμων για την ομάδα των ε, Σοσιαλιστών προτείνω την συνάδελφο Άννα Γκόμες. Ε, και εδώ βεβαίως ισχύει αυτά που είπε και για μένα πριν ο κύριος Φέρμπερ. Πρέπει να διαπιστώσουμε την απαρτία. Βλέπουμε ότι υπάρχει απαρτία πριν περάσουμε στην πληροφορία. Πρέπει, προτείνονται οι υποψήφοι. Πρώτη υποψηφιότητα είναι η υποψηφιότητα των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών. Βεβαίω πρέπει να ρωτήσω αν υπάρχουν άλλε προτάσει, άλλε υποψηφιότητε από τι υπόλοιπε ομάδε. Όχι. Η κυρία Γκόμες είναι παρούσα, την είδα κάπου. Να, εδώ, απέναντί μου ακριβώ. Να ρωτήσω λοιπόν, ε, χρειάζεται μυστική ψηφοφορία. Όχι. Οπότε μπορούμε διαβοή να ψηφίσουμε την κυρία Γκόμες ως πρώτη αντιπρόεδρο της Επιτροπής μας. Συγχαρητήρια κυρία συνάδελφε και παρακαλώ να λάβετε και τη θέση σας. Στον κατάλογο λοιπόν που έχουμε συμφωνήσει έχουμε τον δεύτερο αντιπρόεδρο, δεύτερη υποψηφιότητα. Εδώ η ECR έχει δικαίωμα να προτείνει. Υπάρχουν ε, προτάσεις. Ποιος είναι ο υπεύθυνο, Ναι, παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Εκ μέρους της ECR προτείνω την κυρία Πυρκορούχονεν Λέρνερ. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. Ε, για το τυπικό να ρωτήσω, υπάρχουν άλλες ε, υποψηφιότητες, άλλες προτάσεις. Όχι. Χρειάζεται να κάνουμε μυστική ψηφοφορία. Όχι. Οπότε διαβοής και πάλι να ψηφίσουμε. Η κυρία Πίρκο Ρούχονεν Λέρνερ εκλέγεται λοιπόν ως δεύτερη αντιπρόεδρος. Τώρα, δικαίωμα πρόταση υποψηφιότητα για τον τρίτο αντιπρόεδρο είναι, έχει η Γκουε. Ε, προτάσεις παρακαλώ. Ποιος θα κάνει την πρόταση. Ευχαριστώ. Εκ μέρου τη ε, ΓΚΟΕ προτείνουμε τον κύριο Φάμπιο Ντεμάση. Ε, Προτείνεται λοιπόν ο κύριο Φάμπιο Ντεμάση. Άλλε προτάσει υπάρχουν. Όχι από ό,τι βλέπω. Χρειάζεται να ψηφίσουμε μυστικά. Όχι. Οπότε πάλι διαβοής μπορούμε να εκλέξουμε τον κύριο Φάμπιο. Δημάση. Συγχαρητήρια κύριε συνάδελφε. Και η θέση σας πλέον είναι εδώ μπροστά. Πάμε τώρα στον τέταρτο αντιπρόεδρο. Οι πράσινοι εδώ ε, έχουν το δικαίωμα της ε, πρότασης. Ο κύριος Γκίγκολτ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εξ των Πρασίνων, θα ήθελα να προτείνω την Εύα Ζολή, την σιδηρά κυρία της ομάδας μας. for in... Και πρώην υποψήφια πρόεδρο. Της Γαλλίας. Ωραία, ακούσαμε λοιπόν την ε, πρόταση των Πρασίνων. Υπάρχει Άλλη πρόταση. Υπάρχει ανάγκη για μυστική ψηφοφορία. Όχι. Διαβοήθηση λοιπόν μπορούμε να εκλέξουμε την κυρία Ζολή. meine sehr verehrten Damen und äh, Ωραία. Συνάδελφοι λοιπόν, όπως ε, προτείνει η απόφαση της Ολομέλειας, έχουμε τον πρόεδρο και τέσσερι αντιπροέδρους. Υπάρχουν ε, παρατηρήσεις ή προτάσεις. Παρακαλώ, κύριε συνάδελφε, κύριε Σίμων. Έχουμε συζητήσει εδώ και πολλές εβδομάδες για την σύσταση της Επιτροπής, γι' αυτό θεωρώ ότι θα πρέπει να αποφασίσουμε και έτσι ένα, σε ένα επικοδομητικό τμήμα, ε, πνεύμα συγγνώμη, την, το Προεδρείο και τους Αντιπροέδρους ένα πέμπτο των εκπροσώπων θα πρέπει ίσως να προκύψει από το Άλντε ε, βεβαίως ε, οι εκπρόσωποι θα καθοριστούν από, τη από την συνέλευση των Προέδρων, αλλά θέλω να πω ότι ε, εδώ, αν δούμε, έχουμε πάρα πολλές ομάδες, ε, οπότε ζητούμε από τη συνέλευση των Προέδρων να συζητήσει το θέμα αυτό και να, να διευκολύνει την εκλογή ενό πέμπτου αντιπρόεδρου από την Άλντε. Ε, δεν ξέρω, υπάρχει ε, άλλος που να θέλει το λόγο. Νομίζω σκόπιμο είναι, αν είναι λογικό. Ε, Βεβαίω αυτό πρέπει να εγκριθεί από το Προεδρείο του ε, Κοινοβουλίου. Βεβαίω η απόφαση ε, μιλάει για τέσσερι αντιπροέδρου. Ο κύριο Ζωζάτη. Εκ μέρου του ΕΛΚ θα ήθελα να στηρίξω αυτό το, αυτή την πρόταση. Πρέπει να έχουμε εκπρόσωπο των φιλελεύθερων στο Προεδρείο αυτής της Εξεταστικής Επιτροπής. Ωραία. Για τη διαδικασία νομίζω ότι χρειάζεται πρώτα η έγκριση και μετά χρειάζεται η εκλογή. Θα γίνει αυτό λοιπόν στην ε, πρώτη μας τακτική συνεδρίαση, μετά από τούτην, την καταστατική μας. Υπάρχουν αντιρρήσεις να γράψουμε μια τέτοια επιστολή. Δεν βλέπω κανένα να έχει αντίρρηση. Οπότε η επιθυμία αυτή που εξεφράστηκε από τους σοσιαλιστές και υποστήριχθηκε από το ΕΛΚ μπορεί να γίνει δεκτή από όλους, σωστά. Ωραία. Προτείνω λοιπόν οι φιλελεύθεροι, εφόσον έχουμε την, α, την επιστολή και την πρόταση, να μας, κάνουν, να μας στείλουν την υποψηφιότητά τους. Ολοκληρώσαμε λοιπόν την ε, ημερήσια διάταξη. Βεβαίω έχουμε διάφορε προετοιμασίε από την ε, γραμματεία και μετά προβλέπετε για ενημερωσή σα μετά την καταστατική συνέλευση να γίνει μια συνάντηση των συντονιστών και μετά, σύμφωνα και με το χρονοδιάγραμμα, η πρώτη μας τακτική συνεδρίαση θα γίνει στις 29 Σεπτεμβρίου. Το διαρεύνησε η Γραμματεία. Ξέρετε ότι πολλά μέλη είναι από την Επιτροπή ε, ΛΥΜΠΕ και από την ΕΚΟΝ και αρχές Σεπτεμβρίου και μέσα Σεπτεμβρίου θα γίνουν ακόμη δύο συνεδριάσεις συντονιστών στις οποίες θα αποφασιστεί πώς θα προχωρήσουμε. Η πρόταση της Γραμματείας για την πρώτη συνεδρίαση ε, ήδη το έχουν αποφασίσει δηλαδή, οι ε, συντονιστές ε, θα γίνει, στην πρώτη συνεδρία θα γίνει η ακρόαση των δημοσιογράφων που έχουν δημοσιεύσει τα Panama Papers. Αυτή ήταν η απόφαση που λήφθη για την πρώτη μας τακτική συνεδρία στις 29 Σεπτεμβρίου. Παρατηρήσεις υπάρχουν από αυτού. Δεν βλέπω κανέναν. Οπότε και πάλι να σας ευχαριστήσω θερμά ο στόχος αυτής της ε, Επιτροπής ε, ορίζεται σαφώς από την ε, συνθήκη διαρεύνηση καταγγελόμενων παραβάσεων και περιπτώσεων κακοδιοίκησης κατά την εφαρμογή της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με την νομοποίηση εσόδων από παράνομε δραστηριότητε, φοροαποφυγή και φοροδιαφυγή, δυνάμει του 198 του ιστορικού κανονισμού. Η εντολή αυτή περιλαμβάνει παραλήψεις της Κομισιόν, των αρχών των κρατών μελών, παραλήψεις της Επιτροπής ε, ε, από το Διοντολογικό Κώδικα και των ε, κρατών μελών, τάξη 1 και 2 και συστάσεις για τη μελλοντική νομοθεσία. Και βεβαίως η δυνατότητα να ασκήσουμε κάποια πίεση. Ξέρετε ότι τα μέλη του Κοινοβουλίου, ως μέλη του Κοινοβουλίου μάλλον, ότι τα κράτη-μέλη γενικώ είναι λίγο δυσκίνητα. Ε, ειδικά όταν πρόκειται για ελεγκτικούς μηχανισμούς της ε, Κομισιόν και του Κοινοβουλίου. Πρέπει λοιπόν το εργαλείο αυτό που μας δίνεται τώρα να το χρησιμοποιήσουμε για να ε, πραγματοποιηθούν τα αποτελέσματα των, της σχετικής νομοθεσίας. 8 Ιουνίου λήφθη η απόφαση. 26 Ιουνίου του 2016 δημοσιοποιήθηκε επισήμως. Η εντολή μας λοιπόν χωρίς να έχουμε ζητήσει ή να ζητήσουμε παράταση, θα ολοκληρωθεί τον Ιούνιο του 2017. Αυτό σημαίνει ότι στην Ολομέλεια του, του Ιουνίου του 2017, αν δεν υπάρχουν λόγοι για να ζητήσουμε παράταση, θα πρέπει να ολοκληρώσουμε την εντολή μας. Είναι ένα αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα που βεβαίως ζητά έντονη συμμετοχή από όλους και εγώ ε, δεν ήμουνα μέλος της Επιτροπής για τα φορολογικά θέματα, αλλά ήμουνα ε, παρόν και ελπίζω ότι και εσείς θα είσαστε παρόντες εδώ, έτσι ώστε να μπορέσουμε να ε, προχωρήσουμε τις εργασίες μας με εντατικό τρόπο. Και ως ε, πρόεδρος πάντα πρόσεχα την παρουσία των μελών και σε μια αντιπροσωπεία στην ε, Ασία έρχονταν μόνο όσοι ήταν παρόντες πάντα στις συνεδριάσεις μας. Οπότε θα είμαι αυστηρός. Θα το ελέγχω, θα ελέγχω τις παρουσίες σας, έτσι ώστε να μην έχουν απαιτήσει όσοι δεν ε, παρίσταντο στι συνεδριάσεις όλη τη χρονιά. Ε, αυτά λοιπόν από μένα. Σα ευχαριστώ πολύ για την εμπιστοσύνη. Να ρωτήσω αν υπάρχει κάτι στα διάφορα που να θέλετε να πείτε. Παρακαλώ κύριε Τόιρερ. Ευχαριστώ. Αγαπητοί συνάδελφοι, ξέρω ότι δεν είναι ε, το σωστό σημείο ή ο χρόνος, αλλά είναι γνωστό ότι σε ό,τι αφορά την ε, ε, εργασία θέλουμε να έχουμε, της Επιτροπής θέλουμε να έχουμε έναν συνεισηγητή. Απλώς ήθελα να πω εδώ στους συναδέλφους ότι η Άλντε θα προτείνει για έναν από τους ε, δύο ε, συζητητέ την συνάδελφο Πέτρα Γέζεκ από την Τσεχία. Σα ευχαριστώ. Υπάρχει και η άτυπη συμφωνία ότι οι σοσιαλιστές έχουν δικαίωμα ε, πρόταση εδώ. Προτάσεις υπάρχουν, ναι. Ακόμα ε, δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία, η τυπική. Μόλις την ολοκληρώσουμε θα σας ενημερώσουμε για τον υποψηφιό μας πρόεδρο. Ευχαριστώ κύριε Σίμων. Κατανοώ, κατανοώ. Δεν, ε, δεν υπάρχει λόγος να ρωτήσω κάτι άλλο. Ε, δεν βλέπω άλλο να αναζητά το λόγο. ολοκληρώνεται λοιπόν η συνεδρία. Σας ευχαριστώ όλους για την εμπιστοσύνη σας και σας εύχομαι καλό καλοκαίρι. Καλές διακοπές.